Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Συνεχίζεται η συνεδρίαση. Τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίαση είναι στη διάθεσή σας. Εάν υπάρχουν σχόλια, αλλά δεν υπάρχουν από ό,τι βλέπω, επομένω συγκρίνονται τα πρακτικά. Και σας ευχαριστώ. Έχουμε δύο θέματα να, συνεχίσουμε, να συζητήσουμε σήμερα επί του προϋπολογισμού. Το πρώτο